θεωρηθούν εγκεκριμένα. του τίτλου λοιπόν των ε, ψηφισμάτων των ε, νομοθετημάτων αυτών θα του βρείτε στα πρακτικά τη κυβέρνηση. Ε, σύμφωνα με την κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία, λοιπόν, ελευθερώθηκαν 7 ε, μια νομοθετική πράξη, η οποία δημοσιεύεται και αυτή στα πρακτικά τη σημερινή συνεδρίαση. Και τώρα, λοιπόν, α περάσουμε